νοτροπία που υφίσταται αυτή τη στιγμή στην Συρία. Εμεί φέρουμε μια τεράστια ευθύνη απέναντι στην Συρία και απέναντι στου χριστιανού τη Συρία. Οι χριστιανοί τη Συρία λένε ότι αισθάνονται ότι δεν έχουν κανένα δικαίωμα και ότι εμεί δεν αφουγκραζόμαστε τι ανάγκε του. Και πραγματικά λυπάμαι που είπατε εκπρόσωπο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θέτουν το ζήτημα αυτό πρωταρχική προτεραιότητα. Εγώ νομίζω ότι η εξωτερική μα πολιτική θα πρέπει να βοηθήσει έμπρακτα του χριστιανού τη Συρία και η ίδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να πλαισιώσει το σύστημα αυτό προστασία. Γιατί διαφορετικά οι κοινότητε αυτέ των χριστιανών κινδυνεύουν με εξαφάνιση. Για ένα λεπτό. κυρία On March the 16th. 16 Μαρτίου ολοκληρώνεται ένα έτος από τότε που η Άννα Κάμπελ ε, δολοφονήθηκε από τις τουρκικές δυνάμεις καθώς υπερασπιζόταν ε, την πόλη του Αφρίμ. Ε, πολεμούσε για την κοινωνική δικαιοσύνη, ήταν τόσο δυσαρεστημένη με όλη αυτή την ανθρώπινη δυστυχία που ε, παρατηρούσε, ώστε αποφάσισε να ενώσει τι δυνάμει τη με ε, τι κουρδικέ δυνάμει στην Βόρεια Συρία, που θεωρούσε ότι ήταν η μοναδικ... ο μοναδικό αξιόπιστο ε, φορέα αντιπολίτευση στο καθεστώ του Ασάντ. Εκείνοι άλλαξαν το ρου του πολέμου και τώρα οικοδομούν εκ νέου ε, την ε, τοπική κοινωνία και με τις γυναίκες ε, στο επίκεντρο αυτής της προσπάθειας. Και εγώ ηγήθηκα μιας ειρηνευτικής αποστολής τον περασμένο Μάιο και είδα με τα μάτια μου αυτή την διαδικασία ανοικοδόμησης. Όμως ένα χρόνο το ισορρός της Άννα ακόμα βρίσκεται κάτω από τα συντρίμια και δεν και πρέπει επιτέλους η Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει μια πραγματική απάντηση σε αυτό. Κυρία Λαλόντ, ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, η κατάσταση στη Συρία είναι πολύ πολύ πλοκή... και ιδιαίτερα επίγουσα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αδύναμη με τους Κούρδους συμμάχους της και δεν θα καταφέρει να συμβάλλει στο μέλλον τους αν δεν συνεργαστείτε, το θέλουμε είτε όχι, με αυτόν που ελέγχει το 90% της επικράτησης χώρας, δηλαδή τον Μπασάρα Λασάντα. Και βέβαια αυτό θα πρέπει να γίνει στη συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών και τι μη κυβερνητικέ οργανώσει. Κύριε Πίτροπε, αν θέλουμε πραγματικά να βοηθήσουμε του Σύριου, θα πρέπει να προβλέψουμε την επιστροφή των Σύριων προσφύγων στην Συρία, όπω το ζητάει ο Λίβανο. Μια χώρα η οποία έχει αναλάβει 1,5 εκατομμύρια Σύριου πρόσφυγε στην επικράτειά τη, θα πρέπει είτε μα αρέσει είτε όχι πάλι να συνεργαστούμε και το ζήτημα αυτό με τον Μπασάρα Λασάντ. Επίση, αν θέλουμε να αποφύγουμε το κίνδυνο της εσωτερικής για την εσωτερική ασφάλεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση, που ενδεχομένω να έχουμε μέσω τη της επιστροφής των χιλιάδων τσιχαντιστών που βρίσκονται αυτή τη στιγμή ε, στις φυλακές της Συρίας ή σε άλλες χώρες και πεδεχομένως να έρθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να συνεχίσουν εδώ τις τρομοκρατικές τους επιθέσεις και για να επιλύσουμε τον κίνδυνο αυτό θα πρέπει, να μας αρέσει όχι, να συνεργαστούμε με τη Δαμασκό. Κύριε Επίτροπε, ποιες είναι οι δικές σας οι δράσεις, οι δικές οι προθέσεις προκειμένου η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει δράση λαμβάνοντα υπόψη την πραγματική γεωπολιτική πραγματικότητα που ισχύει στη Συρία. Κύριε Χατζηγεωργίου, ένα λεπτό κύριε πρόεδρε συζητάμε για όγδοη συνεχή χρονιά και για όγδοη φορά το θέμα της συρίας και δεν ξέρω αν η λέξη απόγνωση μπορεί να περιγράψει το τι αισθάνεται ένας ευρωβουλευτής μετά από 8 χρόνια συζητήσεων. αλλά αν η λέξη απόγνωση δεν αντικατοπτρίζει τι αισθανόμαστε εμείς δεν ξέρω ποια λέξη μπορεί να αντικατοπτρίσει τι νιώθουν οι ίδιοι οι σύριοι μισό εκατομμύριο νεκροί ίσως περισσότερους κατά αναλογία από όσου έδωσε οποιοδήποτε κράτος τη Ευρώπη κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου κατά αναλογία. Και αν η Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε Χάν, ίσως δεν έχει μοχλό προς τη Ρωσία ή προς τις Ηνωμένε Πολιτείε, έχει μοχλό απέναντι στην Τουρκία, η οποία ετοιμάζει μια δεύτερη και τρίτη εισβολή μέσα, στη χώρα τη Συρία και δεν ξέρω ποιο νέο αιματοκύλισμα μπορεί να φέρει αυτό να αξιοποιήσετε όποια όπλα δίνει το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο και η ευρωπαϊκή ένωση στα χέρια σας για να προστατεύσετε τον κουρδικό πληθυσμό από μια νέα επίθεση της τουρκίας έναν πληθυσμό που αγωνίστηκε ενάντια στον isis όσο κανένας άλλος. ευχαριστώ. Βουλή των Κοινοτήτων ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι ο Ασάτ θα παραμείνει στην εξουσία. Αυτό είναι ομολογία όχι απλώς αποτυχίας της Βρετανικής πολιτικής, αλλά και ομολογία αποτυχίας της πολιτικής ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ανεφόρον από το 2012 στήριξε την αλλαγή καθεστώτος. Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα είναι συντρίμια. Το Δεκέμβριο το Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και το Βαχρέιν ξανά άνοιξαν τις πρεσβείες τους ε, στη Δαμασκό. Από ό,τι φαίνεται και ο Αραβικός Σύνδεσμος την ξαναδέχθηκε στους κόλπους του. Ποιος βγαίνει ε, νικητής, ε, Ιράν και Ρωσία. Τελείως παράνομα η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστήριξε τους Ισλαμιστές τρομοκράτες και περιθεροποιήθηκε οριστικά. Τώρα θα κάνει την ίδια ε, λάθος κίνηση ακολουθώντας τους Αμερικανούς στη Βενεζουέλα. Θα πρέπει να αναγνωρίσουν το σφάλμα τους οι Ευρωπαίοι και να ε, ε, ξαναρχίσουν διπλωματικές σχέσεις με την νόμιμη κυβέρνηση στη Δαμασκό. Η μελλοντική μετάβαση θα γίνει ερήμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόσο το καλύτερο η Πρόεδρος. Εδώ διακόπτω το κατάλογο στη διαδικασία κάτσε, όπως σας είχα προαναγγείλει, και δίνω το λόγο στον Επίτροπο, κύριε Χάν. σα παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τα αξιότιμα μέλη ε, του Κοινοβουλίου για την πολύ πολύτιμη συζήτηση και τις τόσο χρήσιμες παρεμβάσεις και ανταλλαγή απόψεων. Από τη συζήτηση αυτή συμπεραίνω ότι υπάρχει συναντήληψη. Όλοι θέλουμε να υποστηρίξουμε τους ήρους και ε, θεωρούμε ότι υπάρχει ανάγκη ε, να ε, επιστρέψουν οι άνθρωποι στις αιστείες τους. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να διατηρήσει χωρίς να χαλαρώνει την υποστήριξή της με τους ίδιους όρους εμείς δεν θα δώσουμε νομιμότητα στο καθεστώς, ούτε θα δεχθούμε ξανά στους ε, κόλπους της διεθνούς κοινότητας σε ένα καθεστώς που δεν θα προχωρεί στις διαπραγματεύσεις και δεν θα σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η διάσκεψη των Βρυξελών είναι για το λαό της Συρίας. Θα έχουμε περισσότερους πολίτες, εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών που θα έρθουν να μιλήσουν με υπουργού μας και με διεθνείς ε, οργανώσεις για τους φόβους, τις αγωνίες και τις ανησυχίες για το μέλλον. Τριήμερη θα είναι αυτή η διάσκεψη και θα έχουμε ε, δύο μέρες ακριβώς ε, την ευκαιρία να συναντήσουν οι άνθρωποι αυτοί τους πολιτικούς και όχι μόνο πολιτικούς αλλά και πολίτες, οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών. Θα έχουν την ευκαιρία να γνωριστούν, να συνομιλήσουν, να ανταλλάξουν απόψεις για να δούμε τι μπορεί να γίνει έτσι ώστε να μειωθεί Ε, το πρόβλημα και να αυξηθεί η ανθρωπιστική βοήθεια και η παροχή της. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να συμμετέχουν περισσότερο οι γυναίκες και να ε, προστατεύονται οι πιο ευάλωτοι. Συνεχίσουμε να παρέχουμε τη βοήθεια της επενδύσης και ε, στο εσωτερικό της Συρίας αλλά και εκτός αυτής ιδιαίτερα στις γειτονικές χώρες που φιλοξενούν τους πρόσφυγες και αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα ακόμα ε, για την ε, υποδοχή των σύρων προσφύγων. Θα πρέπει επίσης να δούμε και την πραγματικότητα κατάματα. Ορισμένοι, αν όχι πολλοί σύροι πρόσφυγες, δεν θα επανέλθουν στο προσεχές μέλλον, είτε μας αρέσει είτε όχι θα πρέπει να δούμε πώς θα υποστηρίξουμε τις ε, χώρες που τους υποδέχονται και τους φιλοξενούν για να αντιμετωπίσουν τα συνεχιζόμενα προβλήματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Ολοκληρώνεται η συζήτηση για το θέμα αυτό. Και προχωρούμε στο επόμενο σημείο κατά την ημερήσια διάταξη που είναι η έκθεση του κυρίου Πρέντα, έκθεση 2018 για τη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Το λόγο έχει ο εισηγητής για Τέσσερα λεπτά παρακαλώ. Uh, uh, σας ευχαριστώ Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, να σε ευχαριστήσω για την εργασία σα, για την αδιάλειπτη δέσμευσή σα για την ευρωπαϊκή προοπτική τη uh, Βοσνία Ερζεγοβίνη. Να που φτάσαμε στην τέταρτη και τελευταία έκθεση για την εξέλιξη της χώρας αυτής και για την πορεία της χώρας αυτής προς την Ευρώπη. Από το 2015 και μετά η Βοσνία Ριζαγοβίνη βρισκόταν σε μια ανωδική πορεία, όλο και πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δυστυχώ όμω από το 2017 και μετά βλέπουμε μια επιβράδυνση που με ανησυχεί και ξέρω ότι ανησυχεί και εσάς κύριε Επίτροπε. Από το 2014 και μετά είμαι μόνιμος συγητή ε, για τη Βοσνία Ερζεγοβίνη και έχω ασχοληθεί ιδιαίτερα με το καθεστώς τη δυνάμει υποψηφιότητα τη χώρα αυτή. Μολονότι έχουν καταβληθεί πολλές κοινέ προσπάθειες να έχουμε καταφέρει να πετύχουμε ακόμα τον σημαντικότατο αυτό στόχο και καθότι καθώς πλησίαζαν μάλλον οι γενικές εκλογές 7 Σεπτεμβρίου του 2018, οι παλαιοί δαίμονες, η πολιτική πόλωση, ο διχασμός, ο εθνοτικός αναδύθηκαν πάλι στην επιφάνεια. Μπήκε η χώρα σε μία εκλογική διαμάχη με μια εκλογική νομοθεσία η οποία ήταν θα έλεγα μερική μόνο με πάρα πολλά άρθρα τα οποία είχαν ακυρωθεί από το σταγματικό δικαστήριο αλλά δεν είχαν αντικατασταθεί από την Βουλή. Τέσσερι μήνε και πέντε μέρε μετά τι εκλογέ βρισκόμαστε σήμερα εδώ και οι αρμόδιε αρχέ, από ό,τι φαίνεται, δεν έχουν καταφέρει ακόμα να συσταθούν, ενώ οι μεταρρυθμίσει καθυστερούν όλο και περισσότερο. Πάρα πολλού λόγου θα μπορούσαμε να εκθέσουμε για τι καθυστερήσει αυτέ. Πολυπλοκότητα τη χώρα, το επόμενο παρελθόν τη χώρα, το τραύμα του πολέμου, το ότι δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η εργασία τη συμφιλίωση. Όλα αυτά θα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μα. Από την άλλη όμω, αυτό το οποίο διακυβεύεται αυτή τη στιγμή δεν να καταφέρουμε να ξεπεράσουμε μια νέα κρίση, αλλά το ίδιο το ευρωπαϊκό μέλλον τη χώρα και ουσιαστικά δεν πρέπει να, είναι, να λογοδοτήσουν σε εμά οι αρχηγοί τη Βοσνία Ερζεγοβίνη, αλλά στου ίδιου του πολίτε του. Οι πολίτε τη Βοσνία Ερζεγοβίνη έχουν και αυτή δικαίωμα σε ένα πολιτικό σύστημα το οποίο θα μπορεί να λειτουργεί και δεν θα εισάγει διακρίσει απέναντι σε κανέναν. Θα πρέπει να μπορούν να ζουν με αξιοπρέπεια στη δική του τη χώρα και να μην αναγκάζονται να φεύγουν στο εξωτερικό. Έχουν ανάγκη και έχουν δικαίωμα από μια ανεξάρτητη δικαιοσύνη η οποία θα λειτουργεί χωρίς να υπάρχει παρέμβαση από την εξουσία, την πολιτική. Οι πολίτε τη Βοσνία Ερζεγοβίνη έχουν και αυτοί το δικαίωμα να ζουν σε μια κοινωνία η οποία δεν θα έχει το καρκίνωμα αυτό τη διαφθορά σε κάθε τομέα του δημόσιου βίου χρειάζονται και αυτοί να έχουν μια διοίκηση η οποία θα είναι αποτελεσματική, αποπολιτικοποιημένη, που θα λειτουργεί υπέρ των πολιτών και όχι το αντίστροφο. Χρειάζονται επίση ανεξάρτητα μέσα μαζική ενημέρωση, τα οποία δεν θα εφίστανται πολιτική πίεση. Η προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί πραγματικά να του προσφέρει όλα αυτά. Και αυτό θα έλεγα ότι είναι εφικτό στην πράξη, αρκεί οι πολιτικές ελίτ της χώρας να εγκαταλείψουν αυτά τα μικρά πολιτικά παιχνίδια τους και να σταματήσουν να υποδαβλίζουν το μίσο προ τι άλλε εθνότητε. Έχει έρθει τώρα η κατάλληλη ώρα να λάβουν τι ευθύνε του οι πολιτικοί αρχηγοί και σε όλα τα επίπεδα να δείξουν ότι λαμβάνουν τι ευθύνε του και ότι θέλουν να προωθήσουν πραγματικά τι οικονομικέ και πολιτικέ μεταρρυθμίσει που θα φέρουν τη χώρα πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πέρα από τις απαντήσεις που πρέπει να δώσει η Βοσνία Ερζεγοβίνη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα στοιχεία αυτά θα δώσουν την ευκαιρία στη Βοσνία Ερζεγοβίνη να πάρει το καθεστώς της υποψήφια χώρας και γιατί όχι ακόμα και φέτο. Τέλος, θα ήθελα να τονίσω το πολύ σημαντικό ζήτημα της συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σα ζητώ επιτακτικά κύριε Επίτροπε να καταστήσετε το ζήτημα αυτό μια πολιτική προτεραιότητα στα επόμενα βήματα της ευρωπαϊκής πολιτικής της Βοσνίας Ερεγοβίνης. Σας ευχαριστούμε κύριε Πρέντα. Καλησπέρα σε όλους. Ο Υπουργός ο κύριος Τσάμπα έχει το λόγο εξ ονόματος Συμβουλίου. Κύριε Πρόεδρε, ξέρω μέλη. Είναι μεγάλη χαρά για μένα να είμαι εδώ σήμερα για να συζητήσουμε την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για το 2018 για την Βοσνία Ριζεγοβίνη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον εισηγητή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Κριστιαν Μπρέντα. Αρχικά θα ήθελα να επαναλάβω την ε, προσήλωσή μας στην ε, ταυτότητα της Βοσνίας ραζεγοβινης ως ενιαίας και ακέραιας χώρας κάτι το οποίο σεβόμαστε πλήρως. Μετά τις ε, εκλογές της 7ης ε, Οκτωβρίου ε, και μετά και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του 2018, περιμένουμε από την Βοσνία Ζεγοβίνη να συνεχίσει τις προσπάθειες για τη διαμόρφωση δομών σε όλα τα επίπεδα προς όφελος των πολιτών ούτως ώστε να ε, ολοκληρωθούν οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις από την πλευρά της χώρας. Το 2016 ε, ξεκίνησε η πρώτη διαδικασία, ε, το οποίο δείχνει ακριβώς την μεγάλη σημασία που έχει για την χώρα αυτή η διαδικασία, όμως πρέπει όλο αυτό να μεταφραστεί και σε απτές πράξεις. Χαιρετίζουμε Ω Προεδρία την, το μήνυμα τη Βοσνία Ερζεγοβίνης ε, για την αποφασιστικότητά τη ε, να ακολουθήσει ε, αυτή την άγουσα και στις 29 και 30 Ιανουαρίου υπόθηκε ότι αναγνωρίζουμε και χαιρετίζουμε τις νέες μεταρρυθμίσεις όπως ε, αυτή για τους ειδικού φόρους κατανάλωσης. Αλλά συμμεριζόμαστε ε, τις ανησυχίε σα, ότι έχουμε χάσει πολύ χρόνο ε, σε διασπαστική ρητορική και προεκλογικέ εκστρατείε που έχουν καθυστερήσει σημαντικά τις μεταρρυθμίσεις παραμένουν ε, σημαντικές προτεραιότητες όπου θα πρέπει να επιτευθούν νέα αποτελέσματα σε ό,τι αφορά το κράτος δικαίου, ε, την ε, οικονομία συμπερίληψης, την μεταρρύθμιση του δημοσίου τομέα, την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης και της τρομοκρατίας και την ενίσχυση της συνεργασίας όλων των επιπέδων διακυβέρνησης. Όντως υπάρχει καθυστέρηση σε ό,τι αφορά την ελευθερία του τύπου και χαιρετίζουμε τις προσπάθειες ε, αντιμετώπισης του ζητήματος. Αναφερθήκατε και στο ψήφισμά σας ότι τώρα μετά τις εκλογές πρέπει όλοι οι πολιτικοί ηθήνοντες να αναλάβουν τις ευθύνες τους ε, για το μέλλον αυτού του λαού. Θα πρέπει η εκλογική μεταρρύθμιση να γίνει ε, σε ένα πλαίσιο διαλόγου για να προσεγγίσει τις ευρωπαϊκές αξίες και πρότυπα αυτή η χώρα. Τώρα, η Προεδρία μας θέλει να αποστείλει πρόσθετες ε, ε, επισημάνσεις στη νέα αίτηση προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Βοσνίας Ρεγοβίνης. Θέλουμε να ενθαρρύνουμε τη Βοσνία Ζεγοβίνη να αξιοποιήσει περαιτέρω ε, τον μηχανισμό προτεξιακής βοήθειας και περιμένουμε και ότι θα διατηρήσει η Βοσνία Ζεγοβίνη την προσήλωσή της σε, σε ολόκληρη τη διαδικασία. Υπενθυμίζω ότι κατά την προετοιμασία της έκθεσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, δίδει ιδιαίτερη σημασία στην ε, υλοποίηση της απόφασης ΣΕΝΤΙΤΖΙ G για την ενοποίηση Κροατών, Σέρβων και Βοσνίων και το Συμβούλιο παραλαμβάνει ότι οι αρχές της ισονομίας όλων των πολιτών και της μη διάκρισης θα πρέπει να διασφαλιστεί πλήρως. Συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε την χώρα στις προσπάθειές της ε, να προχωρήσει σε ε, νέες μεταρρυθμίσεις, ε, στην, προσέγγιση, στην προσπάθειά τους να ακολουθήσουν την ευρωπαϊκή άγουσα. Θα υπάρξει και η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής λοιπόν, για την αίτηση της Μασής Ριζογοβίνης. Θα τα δούμε όλα και εκεί. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Ο Επίτροπος Χάντορ έχει το λόγο στο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κύριε Πρόεδρε, Υπουργέ, αξιότιμα μέλη. Καταρχάς θα ήθελα πραγματικά να ευχαριστήσω τον εισηγητή Κρίστιαν Νταν Πρέντα για το ψήφισμα αυτό, την έκθεση για την Βοσνία Ερζεγοβίνη. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω όχι μόνο εσάς αλλά και κάποιους από τους συναδέλφους σας για ε, την ακούραστη ενασχόλησή σας με τη χώρα αυτή και στην χώρα αυτή. Ε, δεν υπάρχουν ε, ακόμα συγκεκριμένα αποτελέσματα, αλλά μοιραζόμαστε την ίδια προσήλωση και το ίδιο ενδιαφέρον να θέσουμε τη χώρα αυτή όχι μόνο προς την ευρωπαϊκή κατεύθυνση αλλά και για να βοηθήσουμε να ε, βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης του λαού στη χώρα αυτή γιατί αυτό μετράει τελικά και αυτό έχει σημασία και θα πρέπει να είναι ο ακούραστος ε, στόχος μας. Το κείμενο είναι ισορροπημένο και σε γενικές γραμμές ευθυγραμμίζεται με την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Βοσνία Ερζεγοβίνη του Απριλίου 2018. Περιγράφει καλά την κατάσταση στη χώρα και τα προβλήματα και τα εκκρεμώντα ζητήματα για την ενταξιακή πορεία της Βοσνίας καλώς Καλωσορίζω την υποστήριξη της προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που περιγράφει η έκθεση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό σε μια κρίσιμη στιγμή για τη χώρα και τους νεοκλαϊγέντες ηγέτες της. Ανέλαβαν κάποιες ε, δεσμεύσεις και έκαναν υποσχέσεις πριν τις εκλογές. Τώρα αυτά θα πρέπει να γίνουν πραγματικότητα. Είδαμε ρητορική, διχαστική και χρειάζεται να δημιουργηθούν δομές για να κυβερνηθεί η χώρα για να ε, φτάσει ε, στο στόχο της που είναι η ευρωπαϊκή ένταξη. Αυτό ήταν και το μήνυμα που έστειλαν ο πρόεδρος Τούσκο, ο πρόεδρος Γιούνκερ, η κυρία Μογκερίνη και εγώ που είχαμε την ευκαιρία να συναντηθούμε με τους ηγέτες της Βρυξέλλες ε, ήταν ε, το πρώτο του ταξίδι στις Βρυξέλλες ε, μετά τις εκλογές ε, και είπαν ότι και οι πολίτες ζητούν την ευρωπαϊκή ένταξη της Βοσνίας Ερζεγοβίνης. Και εμείς θέλουμε πρόοδο ε, προς την Ευρωπαϊκή Ένωση οριστική και μη αναστρέψιμη. Ταυτόχρονα όμως τονίσαμε και στα μέλη ε, της Προεδρίας ότι χρειάζονται ε, συνολικές μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει από άλλες χώρες στην προεκταξιακή του πορεία. Το θέμα δεν είναι να δοθούν μόνο απαντήσεις στις ερωτήσεις μας από το ερωτηματολόγιο Βεβαίως περιμένουμε προσεχώς να δοθούν αυτές οι απαντήσεις, αλλά δεν σταματάει εκεί η ε, υπόθεση. Θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένα αποτελέσματα στη δημόσια διοίκηση, στη δικαστική μεταρρύθμιση, στο κράτο δικαίου, ανθρώπινα δικαιώματα, χρηστή διακυβέρνηση, που να ευθυγραμμίζονται με τι αρχέ και τι αξίε και του κανόνε Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, εκεί θα κρυθεί η νέα Προεδρία και έτσι θα αξιολογήσει την ετοιμότητα ε, τη χώρα αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση για ακόμα μεγαλύτερη πρόοδο και για την ευρωπαϊκή της πορεία. Για πρώτη φορά θα δώσουμε ένα συνολικό δικό χάρτη όταν κάνουν αίτηση η ένταξη ε, προωθούμε και αναβαθμίζουμε την τεχνική μας βοήθεια ε, στο κράτος δικαίου, στα ανθρώπινα δικαιώματα, θεμελιώδη δικαιώματα, και συγκεκριμένα ε, θέματα και περιπτώσεις. Έχουμε διπλασιώσει την χρηματοδοτική βοήθεια μας 80 εκατομμύρια ετησίως για την περίοδο 2017-2020 ε, βοήθεια, όχι δάνεια, για κάποιες στρατηγικές σε θέματα ενεργειακά, περιβαλλοντικά ή ανάπτυξη της υπαίθρου. Ως τμήμα ε, έργων για τη διασύνδεση στην περιοχή. Τέλος, θέλω να τονίσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξακολουθεί να υποστηρίζει τη Βοσνία Ερσεγοβίνη, γιατί πιστεύουμε ότι το μέλλον της είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ταυτόχρονα υπάρχουν προκλήσεις και προβλήματα που πρέπει να λυθούν με τρόπο σοβαρό και χρειάζονται σοβαρές προσπάθειες από τους εκλεγέντες τώρα ηγέτες της χώρας. Εμείς, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, μπορούμε να βοηθήσουμε με καθοδήγηση και βοήθεια, αλλά εκείνοι είναι οι μόνοι που μπορούν να απαντήσουν στις προσδοκίες των πολιτών τους. Ε, στο πλαίσιο αυτό θα μεταβώ στο Σαράγεβο το πιθανότερο τέλη Μαρτίου για να αποτυπώσουμε την πρόοδο που έχει κάνει η κυβέρνηση και να ε, προχωρήσουμε. Αυτό που τώρα έχει σημασία όμως και είναι απαραίτητο και πρέπει να τονίσω ξανά και ξανά είναι ότι όλοι μας λένε στη Βοσνία Ζαγοβίνη ότι είμαστε όλοι υπέρ της ευρωπαϊκής πρόπτικης και πορείας της χώρας. Τι λείπει όμως συνεπής και συνεκτική ε, δράση επιτόπου όπου να συμμετέχουν όλα τα πολιτικά κόμματα και όλες οι εθνότητες, να προχωρούν σε ένα ενωμένο δρόμο, ε, συνεκτικό. Γιατί πάνω από 80% των πολιτών το επιθυμούν αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε κύριε Πίτροπε. Ας ακούσουμε τώρα την άποψη των πολιτικών ομάδων. Δεν μπορούμε να δεχθούμε στη φάση αυτή μπλε κάρτα γιατί έχουμε καθυστερήσει. Εξ του ΕΛΚΑ, η κυρία Σουίτσα έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να ευχαριστήσω τον κύριο Χάν, τον Επίτροπο και να ευχαριστήσω βέβαια και τον εισηγητή μας, τον κύριο Πρέντα. Είδαμε ότι υπάρχει μια γενικότερη τάση της Βοσνίας να έρθει πιο κοντά στην Ευρώπη, αλλά όπως ακούσαμε από την συγκητή επιβραδύνθηκε η Ευρωπαϊκή Προοπτική το 2017-2018. Και τώρα περιμένουμε μετά τις εκλογές να σχηματιστούν οι διάφορες κυβερνήσεις και αρμόδιες εθνικές αρχές, για το συμφέρον λοιπόν του λαού της χώρας αυτής είναι πάρα πολύ σημαντικό να προχωρήσουν οι μεταρρυθμίσεις αυτές που θα φέρουν πιο κοντά τους πολίτες και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς έχουμε επιμήκη σύνορα με την χώρα αυτή. Ενδιαφερόμαστε λοιπόν πάρα πολύ για τη Βοσνία Ερζεγοβίνη ως Κροάτες και ελπίζουμε πραγματικά ότι ο δρόμος αυτός που θα φέρει τη Βοσνία Ερζεγοβίνη προς την Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι σύντομος και γρήγορος. Παράλληλα όμως θα πρέπει να θυμηθούμε και κάποια πράγματα. Έναν εκλογικό νόμο που δεν έχουν, δεν έχουν ακόμα μεταρρυθμίσει και αυτό θα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα και θα αποτελέσει βάση και τι υπόλοιπε μεταρρυθμίσεις που θα πρέπει να λάβουν χώρα. Θα πρέπει επίσης να αποφύγουμε οποιαδήποτε πολιτική εμπλοκή στις εκλογές, πράγμα το οποίο το είδαμε στο παρελθόν και ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν ε, ορισμένοι πολίτες στη Βοσνία Ριζαγοβίνη που δεν έχουν ισότιμα δικαιώματα με τους υπόλοιπους. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει ισότητα δικαιωμάτων στη Βοσνία Ριζαγοβίνη. Οι νέοι πολιτικοί θύνοντε, οι νέοι πολιτικοί αρχηγοί φέρουν μια τεράστια ευθύνη αυτή τη στιγμή. Και ελπίζουμε ειλικρινά ότι θα καταφέρουμε να του κάνουν να αναλάβουν τι ευθύνε του αυτέ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κύριο Φλέκενστάιν και εξ ονόματος του κυρίου Παπαδάκη που ε, αποσιάζει σήμερα για την κολλήτη, θέλω να με ευχαριστήσουμε τον κύριο Πρέντα. Η έκθεση είναι σχεδόν πλήρης, πολύ λεπτομερής και δείχνει και αποτυπώνει την πραγματική κατάσταση όπως τη βλέπουμε και εμείς οι σοσιαλιστές και δημοκράτες. Ο δρόμος προς την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ανοιχτός για τη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι και εμείς οι σοσιαλδημοκράτες θέλουμε η Βοσνία Ριζεγοβίνη να ακολουθήσει αυτό το δρόμο και να το βρει προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ακριβώς επειδή το επιθυμούμε και από συμπάθεια προς τους ανθρώπους στη χώρα θέλω να πω και μερικά επικριτικά λόγια. Επιθυμούμε να γίνουν οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις στη χώρα για να προχωρήσουν με ε, ταχύτερους ρυθμούς και καλύτερους. Η συμφιλίωση δεν έχει ε, προχωρήσει δραστήρια. Παραμένουν ακόμα πολλά διχαστικά και λίγα κοινά στη χώρα αυτή. Ακόμα οι κυβερνώντες δεν κάνουν βήματα για να ξεπεράσουν το διχασμό του παρελθόντος και να τον ενταφιάσουν. Η συμφωνία του Ντέιτον ήταν πάρα πολύ μεγάλος κόπος και εξαιρετική προσπάθεια για να τερματίσει τον πόλεμο. Αλλά προφανέστατα δεν βοηθάει καθόλου να στηθεί ένα ενιαίο κράτος. Γι' αυτό κατά την άποψή μας θα πρέπει από τις Βρυξέλλες να ξεκινήσει μια πρωτοβουλία για ένα δεύτερο Ντέιτον. Όλο και περισσότερο όταν πηγαίνω στη χώρα έχω την εντύπωση ότι όλο και πιο πολλοί άνθρωποι θέλουν τη συμβίωση και οι ε, ε, υπεύθυνοι πολιτικοί υπολείπονται κατά πολύ ε, αρμόδιοι και υπεύθυνοι και στη Βοσνία Ερσεγοβίνη θα λογοδοτήσουν κάποια στιγμή απέναντι στο λαό τους και θα πρέπει να εξηγήσουν γιατί παραμένουν σε αγκυλώσεις εθνικές του παρελθόντος αντί να φέρνουν πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση μια νέα σύγχρονη Βοσνία. Ευχαριστώ πολύ. Εξ του ECR, ο κύριος Μπέλτερ για 1,5 λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Από την περασμένη χρονιά προέκυψαν ε, ενδιαφέρουσε επιστημονικές αναλύσεις στη Βέννη με το, τον τίτλο ε, αμερόληπτο δημοσιολαβητέ ή ανταγωνισμό ε, προ την Ευρωπαϊκή Ένωση, Τουρκία και ο ρόλο τη στα Βαλκάνια. Οι σχέσει μεταξύ Άγκυρα και Σαράγεβο ε, καταδεικνύονται ιδιαίτερω σε αυτή την ανάλυση. Φυσικά υπάρχουν και προσωπικοί και πολιτικοί δεσμοί ε, μεταξύ Αντογάν και Μπέγκοβιτ. Και με διαπίστωση, διαπίστωση αυτή φτάνουμε και στην παράγραφο 14 του, ε, της έκθεσης Φρέντα που μιλά για την ε, επιρροή εξωτερικών δυνάμεων στη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Το ερώτημά μου είναι κατά πόσο αυτή η ανάλυση έχει ληφθεί υπόψη είναι πραγματικός ε, ε, αντικειμενικός διαμεσολαβητή ε, η Τουρκία στα Βαλκάνια. Υπάρχει και η Ένωση των Ευρωπαίων Βαλκανικών Δημοκρατών και με ιδιαίτερα συμφέροντα και πολύ μεγάλη σημασία. Πρέπει να υπάρχει σαφής και άμεση ευρωπαϊκή απάντηση γιατί αυξάνονται και τροφοδοτούνται οι εντάσεις μεταξύ των εθνικών ομάδων. Για τους φιλελεύθερους, ο κύριος Ράντος έχει το λόγο για δύο λεπτά, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, ε, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον κύριο Πρέντα για την καλή συνεργασία και για την καλή του έκθεση. Είναι η τελευταία έκθεση στην παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο και είχαμε την ευκαιρία πέντε χρόνια τώρα να δούμε ε, και να μετρήσουμε αν ήταν μεγάλη ή μικρή η μικρη η προοδο της Βοσνίας Ερζεγοβίνης προς την Ευρώπη. Τώρα έχουμε μηχανισμούς συντονιστικούς ε, έχουν καταθέσει και την αίτησή τους. Έχουμε ένα πρώτο ερωτηματολόγιο που ε, απαντήθηκε και επίσης έχουμε διάφορες τομεακές στρατηγικές. Αλλά ποιο είναι το βασικό πρόβλημα της χώρας. Είναι ότι δεν λειτουργεί η χώρα. Ε, με εσωτερικούς διχασμούς, με βάση εθνοτικές γραμμές παραμένουν τα προβλήματα. Και μπορούμε να πούμε σχεδόν ότι αυτό είναι υποκειμενικό ε, το αν λειτουργεί ή όχι η χώρα, αλλά η κατάσταση είναι δύσκολη και άσχημη. Ε, δεν υπάρχει ε, σταθερότητα και ασφάλεια στη χώρα. Ε, ίσως είναι αυτή λιγότερη από ότι πριν από πέντε χρόνια. Εμείς μπορεί να έχουμε θεσμικά όργανα και πολιτικούς θεσμούς, αλλά καταλήγουμε ότι είναι προτεραιότητα η Βοσνία, η Ζεγοβίνη και τα άλλα κράτη της περιοχής να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτός είναι ο σκοπός και είναι καλός ο στόχος. Ε, ε, η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι επίση πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ καλή, παρόλο που ορισμένα πράγματα θα έπρεπε να είναι πιο συνεπή. Γιατί ε, ανάμεσα στην παρουσίαση, στην περιγραφή και στα συμπεράσματα υπάρχει αντιστοιχία. Τι θέλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτά που έχουμε κάνει τα τελευταία πέντε χρόνια δεν αρκούν. Θέλουμε η Επιτροπή να εμπλακεί περισσότερο, να υπάρχει μεγαλύτερη, περισσότερη δουλειά και πολιτική για του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου, έτσι ώστε να βοηθήσουμε τη Βοσνία Ριζεγοβίνη με ταχεία πορεία, με ταχεία βήματα να πάει προς τη δική της ασφάλεια και σταθερότητα. Ο κύριος Κόχλιτσεκ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Βοσνία ριζαγοβινη είναι μια πρώην χώρα της πρώην Ιουκοσλαβίας με πολύ μεγάλη πολυπλοκότητα όσον αφορά την εθνοτική της διαμόρφωση. Πολλές οι διαφορετικές εθνικότητες αλλά και μια έντονη θρησκευτική δομή. Έχουμε πολλούς μουσουλμάνους, έχουμε ορθόδοξες εκκλησίες στην Ήπεθρο, έχουμε και τον καθολικό πληθυσμό στα βόρεια ανατολικά. Έχουμε τους Σέρβους, τους Βόσνους, Μουσουλμάνους και τους Κροάτες που μιλάνε τρεις διαφορετικές διαλέκτους μιας κοινή όμως γλώσσας. Μετά τον Φρικαλαίο πόλεμο, τον οποίο υποστήριξαν και ξένες δυνάμεις, έχουμε δύο οντότητες μία στα βόρεια τη Σερβική Δημοκρατία τη Βοσνία Ερζεγοβίνη, τη Ρεπούμπλικα Σρέψκα και μία ακόμα αντότητα την Ομοσπονδία Βοσνία Ερζεγοβίνη. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να αλλάξει τώρα την δομή αυτή τη χώρα, μολονότι προβλέπεται κάτι τελώ διαφορετικό συμφωνία του Ντέιτον και μολονότι δεν το θέλει αυτό ούτε καν ο λαό τη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Δεν νομίζω λοιπόν ότι μπορούμε εμεί ω εξωτερικοί παράγοντε στα πλαίσια τη προσχώρηση να επιβάλλουμε προποθέσει οι οποίε προβλέπουν την αλλαγή της ε, εθνοτικής ε, διάρθρωσης της χώρας αυτής. Ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή έντονες διασυνδέσεις μεταξύ της Βοσνίας Ερζαγοβίνης και άλλων όμορων χωρών, ιδίως όσον αφορά τις οδικές και τις σιδηροδρομικές μεταφορές. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει εμείς να ευνοήσουμε και να προωθήσουμε μια καλύτερη συνύπαρξη μεταξύ των τριών αυτών συστατικών εθνοτήτων και συνεχίσουμε να επικρίνουμε τους αρχηγούς Τη Βοσνία Ερζεγοβίνη, του πολιτικού αρχηγού, αν αγνοούμε τα, τα εγκλήματα πολέμου τα οποία διέπραξαν οι διάφορες στατικές εθνότητες και βέβαια και το σημαντικότατο έγκλημα στην Σεμπρένιτσα, τότε τα πράγματα δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να βελτιωθούν. Εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει ως Ευρωπαϊκή Ένωση να συμβάλλουμε περισσότερο στο κοινωνικό τομέα, στο τομέα της κατάρτισης και της εκπαίδευσης και να μην επιβάλλουμε όλο και νέες απαιτήσει στη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Για τους πράσινους, ο κύριο Σόλτες, δύο λεπτά. Η Βοσνία Ζεγοβίνη είναι μια πολύ αντιφαντική χώρα. Με πολλά στοιχεία που τη συνδέουν. Κατά τη διάρκεια της ιστορίας της έγιναν πολλές αλλαγές Καλό είναι να διαβάσετε τη γέφυρα στο Δρίνα του Ιβάντριτς. Θα σας βοηθήσει να καταλάβετε την τέχνη της συνύπαρξης στη χώρα αυτή. Η Βοσνία Ζεγοβίνη ξεκίνησε το δρόμο προς την ευρωπαϊκή εμνοποίηση. Ο δρόμος αυτός δεν είναι εύκολος και έχει πολλά εμπόδια. Προφανώς όλοι θέλουμε τα κράτη των Δυτικών Βαλκανίων να γίνουν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά οι χώρες αυτές πρέπει να περάσουν μία διαδικασία μεταρρυθμίσεων, αλλαγών, προσαρμογών που απαιτεί ο δρόμος αυτός. Η έκθεση που έχουμε μπροστά μας σήμερα περιλαμβάνει πολλές απόψεις. Αυτό που ωστόσο είναι κοινό σε όλες τις απόψεις είναι ότι Πολλά πρέπει να γίνουν ακόμα. Αντιμετώπιση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος, μεταρρύθμιση του δικαστικού, προστασία των μειονοτήτων, περιβαλλοντικές προκλήσεις πολλές, ελευθερία του τύπου, η παιδεία, θα μπορούσα να πω και κάτι ακόμα. Πρέπει όταν μιλάμε για τη χώρα να σκεφτόμαστε το λαό της Βοσνίας ε, Μια ισχυρή Βοσνία είναι ισχυρή Ευρώπη. Ο κύριος Έφεριτζ για το EFDD, δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Όταν ακούω τις συζητήσεις και εκθέσεις για την ένταξη νέων χωρών ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θυμάμαι το Star Trek, το ταξίδι στα αστέρια. Θυμάστε την ταινία, το Μπόργκ που έλεγε ότι ε, θέλουμε μέσα στο πλοίο της, ε, μέσα στο διασμόπλαιο να συνυπάρχουν όλες οι, εθνικοί, όλες οι, οι φυλές, όλα τα είδη. Ε, ο καθένας ζητάει κάτι δικό του από την ε, συγκεκριμένη θερμοκρασία μέχρι τον ειδικό φωτισμό. Δημιουργούμε χώρους που βοηθούν τον καθένα, αλλά αν δούμε την πραγματικότητα θα καταλάβουμε ότι έχουμε μία κατάσταση όπου η αυτοκρατορία της Ένωσης θέλει να φέρει τους πάντες μέσα, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τις πιθανές μορφές βίας, το εμπόριο, την, ε, τις συγκρούσεις. Όταν συνεχίζεται να επεκτείνεται προς την κατεύθυνση αυτή σε πολύ ευαίσθητους χώρους όπως τα Βαλκάνια, προσέξτε το. Πρέπει να προσέχετε ιδιαίτερα όταν αν εξετάζετε από πού θα προέρχονται τα χρήματα για την ενσωμάτωση των ολοένα και φτωχότερων χωρών στην Ένωση. Ξεχνάτε στη φάση αυτή ότι σε κάποια στιγμή στο εγγύς μέλος θα χρειάζεστε χρήματα. Διότι αν δεν υπάρξει μια συμφωνία με το Brexit θα έχετε πολύ, μεγάλο, πολύ μεγάλη τρύπα στον προϋπολογισμό σας. Μην προσφέρετε πολλά καρότα σε κόσμο πριν προσπαθήσετε να φτιάξετε έναν καινούργιο κόσμο για σας. Ο κύριος Μποτζεγκέτσιο για το ΙΕΝΕΦ. E Ένα λεπτό. Χωρίς μικρόφωνο. Η κατάσταση στη Βοσνία όπως ανακύπτει ε, ειλικρινά και με σαφήνεια δείχνει τις μεγάλες δυσκολίες που υπάρχουν σε αυτή την ε, πορεία προσχώρησης προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για μια ε, χώρα που έχει κάνει πολύ μικρή πρόοδο από τότε που άνοιξε η διαδικασία και αναρωτιόμαστε κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση με τους οικονομικούς της περιορισμούς έκανε ότι ήταν αναγκαίο και ήταν στο ύψος των περιστάσεων για να ηγηθεί αυτού του λαού. Πέρα από την ιστορία που είναι γνωστή σε όλους. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε και την γεωπολιτική θέση της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης και τους κινδύνους που υπάρχουν. Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος διείσδησης ξένων μαχητών. Αυτός είναι μεγάλος κίνδυνος. Ο κύριος Κούκαν για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή γιατί ασχολήθηκε με αυτό το θέμα εδώ και πέντε χρόνια. Δυστυχώς οι τελευταίοι μήνες δεν οδήγησαν σε μεγάλη πρόοδο της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης για να προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι ηγέτες ε, θέλουν στην ουσία να επανδρώσουν τα ε, Υπουργεία και τα, σώμα, διάφορα σώματα και αυτό μέσα στα πλαίσια της ε, διαδικασίας για μελλοντική προσχώρηση. Υπάρχει επίγον ζήτημα αντιμετώπισης αναθεωρήσεων για την ε, πλήρη εφαρμογή κράτους δικαίου. Πρόκειται για ε, στόχους για το μέλλον. Προσπαθούμε να συνδράμουμε και ως προς τον εκλογικό νόμο και την αναθεώρηση του συντάγματος. Ελπίζω η Βοσνία και η Ερζεγοβίνη να δεχτούν αυτή τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, ε, ε, θεωρούμε ότι θα πρέπει να καταπολεμηθεί η μισαλοδοξία και η ρητονική μίσους και αυτό αφορά και το εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο εντάσσει αυτά τα ζητήματα προς αντιμετώπιση. Πιστεύω ότι υπάρχει η ευρωπαϊκή προοπτική της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης και θα δώσει, ότι θα δώσει μεγάλη μάχη για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος Πίτσουλα έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Από το 2015 και μετά συζητούμε τις ε, ετήσιες εκθέσεις και όχι μια εκθέση πρόοδου. Είναι γεγονός ότι δεν υπάρχει πρόοδος. Ίσα ίσα διαπιστώνουμε παλινοδίες. Μιλάμε για οικονομικές πολιτικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις και δυστυχώς δεν υπάρχουν καλές σχέσεις, θεσμικές σχέσεις και συζητήθηκε πέρσι και ο εκλογικός νόμος, αλλά δυστυχώς ε, δεν ευθυγραμμίστηκε με βάση την απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου. Και μετά τις εκλογές έγινε λόγος για επικουρικότητα, φεντεραλισμό και ό,τι κάναμε μετά το 2013 θα πρέπει να ολοκληρωθεί αυτή η μετάβαση έτσι ώστε όλοι να είναι ίσοι στη χώρα αυτή. Δυστυχώς, το φετινό έγγραφο δεν υπάρχουν αυτά τα στοιχεία και είναι μια μεγάλη παλινοδία. αυτό δεν μπορώ να υποστηρίξω, ή να υποστηρίξω την έκθεση αυτή. Η κυρία Τόμασιτς, η Ευρωπαϊκή Ένωση ακολούθησε την ίδια θέση που είχε ακολουθήσει και στο παρελθόν και η εκλογική προεκλογική εκστρατεία ακολούθησε την ίδια ιστορική πορεία του παρελθόντος. Οι Βρυξέλλες δεν κατανοούν την κατάσταση. Το θέμα της εθνικής ταυτότητας είναι πολύ σημαντικό και δεν θα σταματήσει επειδή μερικοί απλώς το θέλουν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βοήθησε για να δημιουργηθεί αυτή η πολύ όμορφη χώρα όπου και γεννήθηκα. Αλλά δυστυχώς είναι ένας δοκιμαστικός σωλήνας για τη διεθνή κοινότητα. Οι Κροάτες επέλεξαν τον εκπρόσωπό τους με μια διαδικασία που δεν ήταν καθόλου διαφανής και υπάρχει θέμα πολιτικής ταυτότητας. Πάντα ευρωπαϊστής ο συνάδελφος Πρέντα. Μια Ευρώπη που ούτε δούλεψε ούτε θα δουλέψει. Κάνει μια προσπάθεια να μετατρέψει τη Βοσνία Ζεγοβίνη σε ένα μεταεθνικό κράτος και να μην αναγνωρίσει τις τρεις εθνικές ομάδες με συνταγματικά δικαιώματα η καθεμία. Η στρατηγική αυτή μπορεί να οδηγήσει μόνο στην κυριαρχία του, μουσουλ, του πλειοψηφούντος μουσουλμανικού πληθυσμού και μια χρόνια αστάθεια. Η καταδίκη του εθνικιστικού λόγου από πλευρά του είναι καταδίκη έμεσα της Ρεπούμπλικα Σέρψκα. Η Ένωση πρέπει να σταματήσει να αγωνίζεται για την καταστροφή των εθνικών ταυτονοτήτων. Η ένταξη της Βοσνίας στην Ευρώπη σημαίνει άρνηση της Ευρώπης των εθνών, άρνηση των εθνικών ταυτοτήτων. Αυτή η Ευρώπη τέλειωσε. Δεν υπήρξε ποτέ άλλωστε. Πρέπει να δημιουργηθεί η Ευρώπη της συνεργασίας μεταξύ εθνών. Η κυρία Ζόφκο, 1,5 λεπτό. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, χαιρετίζω τη συμφωνία που επιτεύχθηκε την Κυριακή μεταξύ των επικεφαλής των ε, Σέρβων και των ε, Κροάτων στο Μόσταρ κάτι που χαιρετίστε και εσείς και η κυρία Μογκερίνη μετά τις εκλογές. Οι ηγέτες ε, των βοσνιακών ομάδων της, της μουσουλμανικής βοσνιακής ομάδας πρέπει να μετάσχουν τη σύμφωνη αυτή για να αποφευχθεί μια νέα ανάφλεξη ιδίως στο Μπίχατς. Είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι βλέπουμε πως ο κύριος Κόπνιτς, επικεφαλής των μουσουλμάνων Βόσνιων, αρνείται, χρησιμοποιεί μάλλον μη συνταγματικές μεθόδους για την προσέγγιση του ζητήματος. Πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι συγκειτονικές χώρες να παρέμβουν προς όφελος της ειρήνης. Το ίδιο πρέπει να κάνουμε και εμείς από την ε, από πλευράς για να περάσουμε από την περίοδο του Dayton στην περίοδο των Βρυξελών. Η κυρία Φαγιόν. Δεν ξέρω για πόση πρόοδο μπορούμε να μιλήσουμε στη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Αν ένα κράτος ε, ε, ε, ήθελε ποτέ βοήθεια από μας για να προοδεύσει, είναι η Βοσνία Ζεγοβίνη σήμερα. Η επίσκεψη τριών μελών της Προεδρίας της χώρας της Βρυξέλλες μας δίνει ελπίδα ότι μπορεί να επιτευχθεί μια συνενετική λύση στην πορεία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει πάντα τα λόγια να ακολουθούνται από έργα. Αυτό, εάν δεν γίνει, δεν μπορεί να βοηθήσει. Επίσης, η Βοσνία Ζεγοβίνη πρέπει με βάση τις ε, κατευθύνσεις γραμμές της Κομισιόν να διαμορφώσει την ε, ε, κυβέρνησή της και να αναλάβει και νέες πρωτοβουλίες. Να μην ξεχάσουμε παρά το ότι επίκενται εκλογές τη Βοσνία Ζεγοβίνη, παρά το ότι δεν επιφέρει κανένα μικροκομιτικό όφελος για κανένα οι ηγέτες πρέπει να κληθούν να ξεπεράσουν τις ε, διαφωνίες τους. Ε, η κυρία Πετήρ, κύριοι επίτροπε συνάδελφοι, ευχαριστώ τον συνάδελφο Πρέντα γιατί αποδέχθηκε μερικές από τις προτάσεις μου, τις οποίες συζητάμε σήμερα. Αλλά εάν μιλάμε για την κατάσταση στην ε, Βοσνία Ζεγοβίνη, φαίνεται ότι παρά όλες τις προσπάθειες που κάνουμε δεν κινείται τίποτα ουσιοδός και ενώ εμείς ως κοινοβούλιο θέλαμε να αλλάξει ο εκλογικός νόμος στην Βοσνία τελικά προέκυψε μια κατάσταση όπου οι Κροάτες ε, δεν μπόρεσαν να εκλέξουν τους εκπροσώπους τους. Υφίστανται διακρίσεις οι Κροάτες στη Βοσνία Ζεγοβίνη. Η θέση της Βοσνίας Ζεγοβίνης είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το θέλω με όλη μου την καρδιά. Αλλά πρώτα απ' όλα η Βοσνία Ζεγοβίνη πρέπει να ε, τηρεί τη συνταγματική νομιμότητα. Πρέπει να γίνουν οι αναγκαίες αλλαγές. Εφιστώ την προσοχή όλων μας στην ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος στη Βοσνία Ζεγοβίνη Έχουμε ένα διελιστήριο στο Μπόσενσκι Μπρότ, το οποίο πρέπει να λειτουργεί με βάση ε, τις αναγκαίες προδιαγραφές. Μέχρι να γίνει αυτό, δυστυχώς θα εξακολουθεί να βλάπτει το περιβάλλον. Επιπλέον, εφαρμόστε τους κανόνες. Αυτή, αυτή είναι η χρυσή ε, συνταγή. Επίσης η κατάσταση ασφάλειας ε, είναι επισφαλής. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα. Ο κύριος Βάιντεν Χόλτσερ, ένα λεπτό. Έχουν περάσει 20 χρόνια μετά το Ντέιτον. Παρόλα αυτά η Βοσνία Σεγοβίνη δεν έχει ξεπεράσει ακόμη τις επιπτώσεις του πολέμου. Γίνονται πολλές εκκλήσεις υπερβολικές. Γιατί κανείς μετά δεν ε, τις υλοποιεί. Υπάρχουν αυτές οι εντάσεις μεταξύ εθνοτήτων και αυτό δημιουργεί απόγνωση και παντού φαίνεται και εξωτερική επίδραση. Έχει γίνει ε, μπάλα ενό διεθνού παιχνίδιου η Βοσνία Ζεγοβίνη. Υπάρχει τρόπο να ξεφύγουμε αυτό το δίλημα και να δώσουμε μια ευρωπαϊκή προοπτική. Για να γίνει αυτό πρέπει να γίνουν όμω πολύ περισσότερα από ότι να το συζητάμε μόνο μια χρονιά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Χρειάζεται μια νέα δυναμική, η οποία από εμά πρέπει να ξεκινήσει. Οι νέοι και πρώτα απ' όλα, οι νέοι κυρίω ε, και γενικότερο πληθυσμό έδειξαν ότι με τι διαδηλώσει ε, ε, το επιδιώκουν. Μία νέα ε, φοιτήτρια το λέει. Για τη δική μας γενιά δεν μας ενδιαφέρει η εθνικότητα και οι θρησκευτικέ πεπιθήσεις του καθενός, αλλά το πώς να περνάμε καλά μαζί. Ευχαριστώ πολύ. Τελευταία παρέμβαση μέσω της διαδικασίας του Catch the Eye θα ακούσουμε κάποιους συναδέλφους. Παρακαλώ όλοι να είστε συνοπτικότατοι. Σδογεύσκη, ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Πριν 25 χρόνια ήμουν στο Σαράγεβο συνοδεύοντας μία οργάνωση που παρέδιδε ανθρωπιστική βοήθεια κατά τη διάρκεια της πολιορκίας της πόλης. Πρόσφατα ξαναπήγα με επίσκεψη σε αποστολή του Κοινοβουλίου για θέματα ασφάλειας. Ήλπιζα ότι η κατάσταση δεν θα επαν... πριν από 25 χρόνια δεν θα ξανά συνέβαινε. Δυστυχώς υπάρχουν πολλές απειλές και η κατάσταση είναι εξαιρετικά λεπτή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποίησε, έκανε, κατέβαλε προσπάθειες οι οποίες όμως δεν λειτουργούν πλέον. Πρέπει να ξεπεράσουμε την προσέγγιση αυτή. Δεν θα μας βοηθήσει να λύσουμε την εσωτερική κρίση στην χώρα. Πρέπει να έχουμε σαφήνεια στα μηνύματά μας. Παρακαλώ. Ο κύριος Ρόντε. Ο κύριος Γιάκοβτσιτς. Για ένα λεπτό. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η κατάσταση βρίσκεται σε ένα αδιέξοδο στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη. Έχω παρακολουθήσει την κατάσταση εδώ και δεκαετίες. Ξέρω ακριβώς τι συμβαίνει εκεί. Οι πολιτικοί φέρουν την ευθύνη που δυστυχώς δεν είναι στο ύψος των περιστάσεων, δεν ξέρουν τις ανάγκες των πολιτών. Αλλά θα ήθελα να πω ότι οι θρησκευτικοί ηγέτες είναι λίγο πιο προοδευτικοί από τους πολιτικούς. Αυτό μας δίνει κάποια ελπίδα και ο κύριος Χαν έχει κάνει μεγάλες προσπάθειες έτσι ώστε να προσεγγίσει τη Βοσνία και Ερσεγοβίνη και ένα άλλο θέμα είναι οι μετανάστες στη ε, Βοσνία Ερζεγοβίνη. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στηρίζω την έκθεση του συναδέλφου Πρέντα. Είναι πολύ ισορροπημένη και ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Είμαι πεπισμένος, κύριε Επίτροπε, ότι όπως και πριν θα πρέπει με υπομονή να προσφέρουμε ένα ευρωπαϊκό μέλλον στις βαλκανικές χώρες. Και ναι μεν δεν έχουν γίνει επιτυχείς μεταρρυθμίσεις ε, μέχρι τώρα, αλλά δεν πρέπει να εγκαταλείψουμε τη Βοσνία Ζεγοβίνη παρόλα αυτά. Θα ήταν μεγάλο γεωπολιτικό λάθος. Και ε, το κενό αυτό θα το εκμεταλλευόταν η Ρωσία η οποία έχει πολύ καλή επικοινωνιακή πολιτική σε αυτή την περιοχή τώρα τελευταία. Πρέπει λοιπόν να παρακαλέσω να δούμε τη γεωπολιτική διάσταση. Και με υπομονή, επαναλαμβάνω, να επιδιώξουμε να βοηθήσουμε τη Βοσνία Ζεγοβίνη να εφαρμόσει τις μεταρρυθμίσεις που θα την πλησιάσουν στην Ένωση. Ούτω ώστε να μπορέσει να γίνει υποψήφια χώρα. Αν δεν το κάνουμε, η Ρωσία αλλά και η Τουρκία θα τα κάνουν όλα αυτά. Ο κύριος Ζαγιανόπουλο, ένα λεπτό. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Ποιοι άναψαν τους εθνικισμούς στη Βοσνία και αλλού για να διαλύσουν τη Γιουγκοσλαβία, το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η κατάσταση στη Βοσνία συνεχίζει να είναι από τις τελευταίες εκκρεμότητες για την ευρωατλαντική ενσωμάτωση των Δυτικών Βαλκανίων εν μέσω των ανταγωνισμών Αμερικάνων, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Ρωσία και την Κίνα. Οι εθνικισμοί που καλλιεργήθηκαν δεν λένε να κοπάσουν, πυροδοτούν συγκρούσεις, αλλάζουν 20 χρόνια μετά σύνορο όπω τώρα με το Κόσοβο και την Σερβία ανοίγοντα την όρεξη και σε άλλου που διεκδικούν αλλαγέ συνόρων όπω την τουρκία. η επέσχυντη νατοϊκή σκοπή συμφωνία των πρεσπών τσίπρα και ζαεφ προβάλλεται σαν παράδειγμα διευθέτησης όχι για επίλυση διαφορών αλλά για την υπερίσχυση των εμπεριαλιστικών συμφερόντων στα κρίσιμα βαλκάνια. παράδειγμα η μετατροπή και πάλι τις τελευταίες μέρες του λιμανιού της θεσσαλονίκης σε νατοϊκή βάση κάνοντα την δυνητικό στρατιωτικό στόχο των αντίπαλων συνασπισμών που διαψεύδει το μύθο του σύριζα περί σταθερότητας με νατο και ευρωπαϊκή ένωση. ασφάλεια ειρήνη και φιλία των λαών στα βαλκάνια σημαίνει ένα πράγμα να φύγουν το νατο οι αμερικάνοι και η ευρωπαϊκή ένωση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σελίμοβιτς. Έχετε ζητήσει το λόγο, έτσι δεν είναι. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Επίτροπε. Ευχαριστώ που εργάζεστε με τον ίδιο ρυθμό, όχι μόνο στη Βοσνία Ζεγοβίνη, αλλά και ευρύτερα στην περιοχή. Εντυπωσιακό το επίτευγμά σα. Ναι, συμφωνώ με τον εισηγητή. Ο ρυθμό των μεταρρυθμίσεων έχει επιβραδυνθεί από την προεκλογική περίοδο. Ακόμη περιμένουμε να σχηματιστεί κυβέρνηση. Δεν υπάρχει επίσημη συνεργασία με το Κοινοβούλιο και το κράτο δικαίου δεν έχει βελτιωθεί όπω τα ελπίζαμε. Αλλά υπάρχουν ενθαρρυντικά σήματα και βράχη πρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Βράχη πρόθεσμα, καλύτερη οικονομική διακυβέρνηση για παράδειγμα ενθαρρυντικά αποτελέσματα στις ε, αυτοδιοικητικές εκλογές. Η κατάσταση με την τρομοκρατία έχει βελτιωθεί. Και είδαμε τους τρεις προέδρους που ήρθαν εδώ και συνεργάστηκαν. Για πρώτη φορά τους είδα να συνεργάζονται. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να διατηρηθεί ο ρυθμός της ευρωπαϊκής τους προοπτικής. Γιατί δίνει μια προοπτική στη χώρα. Και είναι συνδετική ύλη για να πιάσουν οι μεταρρυθμίσεις. Ευχαριστώ ο κύριος Μαριάς. Ένα λεπτό. Presidente. Ο ανταγωνισμό Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσία στα Βαλκάνια οξύνει τι αντιθέσει. Και βεβαίω τα προβλήματα που δεν μπόρεσε να λύσει τον Ντέιτον, προβλήματα που έχουν σχέση με την ειρηνική συνύπαρξη των εθνοτήτων και των μειονοτήτων στη Βοσνία εντείνονται είναι βέβαιο ότι πρέπει να επαναλάβουμε αυτά που είπαμε και το 2017 σε αυτή την αίθουσα ότι θα πρέπει να υπάρξει δίκαιη αντιμετώπιση των μειονοτήτων μέσα στην βοσνία ερζεγοβίνη ότι οφείλει η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει τα τεράστια προβλήματα που υπάρχουν σε σχέση με τη διαφθορά το οργανωμένο έγκλημα να υπάρξει προστασία ιδίως των ρωμά να υπάρξει εφαρμογή του κράτους δικαίου αξιοκρατία στη δημόσια διοίκηση και γενικότερα προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. θεωρώ λοιπόν ότι όλα αυτά τα οποία είχαμε πει και παλαιότερα δεν έχουν μπορέσει να επιληθούν στην πορεία της βοσνίας ερζεγοβίνης προς την ευρωπαϊκή ένωση ένα εγχείρημα το οποίο φαίνεται ότι δεν μπορεί να επιτευχθεί. ευχαριστώ. Να τονίσω το εξή. Κύριε Επίτροπε, η ασφάλεια και η σταθερότητα στη Βοσνία Ζεγοβίνη είναι κλειδί για την ασφάλεια και τη σταθερότητα ολόκληρη τη Ένωση. Δεν μπορούμε να επιδιώκουμε πολιτική σταθερότητα ε, στην Βοσνία Ζεγοβίνη, αν μία από τι τρει κοινότητε δεν μπορεί να συμμετάσχει στη διαδικασία λήψη αποφάσεων στου θεσμού τη Βοσνία Ζεγοβίνη και να εκλέγει του εκπροσώπου τη. Πρέπει να αλλάξει ο εκλογικό νόμο. Το είπαν και άλλοι εκπρόσωποι πριν από μένα. Να μιλήσω λοιπόν για κάτι άλλο που ίσως δεν τονίστηκε επαρκώς. Είναι η δική μας επιρροή στην Βοσνία Ζεγοβίνη ή η συμμετοχή της Ένωσης στα αναπτυξιακά προγράμματα και διαδικασίες στη χώρα αυτή. Ας αναρωτηθούμε πόσα προγράμματα έχουμε χρηματοδοτήσει μέσω του ΕΦΣΥ στη Βοσνία Ζεγοβίνη. Η απάντηση είναι κανένα. Πόσο έχουμε χρησιμοποιήσει την προενταξιακή βοήθεια. Προσπαθήσαμε να προωθήσουμε κάποια άλλα προγράμματα για να βοηθήσουμε τη χώρα να ενταχθεί στην Ένωση. Τι κάναμε για να ε, οργανώσουμε διάφορα σεμινάρια.